Sorry for that. I was convinced that you were in the middle of working process. Συγγνώμη, νόμιζα ότι θα είχατε αρχίσει. Λυπάμαι που σας έκανα να περιμένετε. Τέλος πάντων. Έγινε μία παρεξήγηση, ας τη θεωρήσουμε μία από τις παρεξηγήσεις. Να αρχίσουμε τώρα με το η συμφωνία πλαίσιο Να αρχίσουμε μια και περιμένουμε, περιμένετε το σύνορα. Λοιπόν, με το Βιετνάμ να αρχίσουμε τότε, με την κυρία Λοχμπίλερ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και την έκθεσή μου την έχω μοιράσει ως εξής τονίζουμε την επιθυμία μας ε, να έχουμε πιο ουσιαστικές ε, σχέσεις ε, με το Βιετνάμ και επίσης καταθέτουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση στις ε, εμπορικές μας σχέσεις, ε, να υπάρχει σωστή και χρηστή διαχείριση, αντιμετώπιση της διαφθοράς, ε, βιοπικιλότητα, προστασία του κλίματος. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες σχετικά με τις διεθνείς προδιαγραφές εργασίες, τα δικαιώματα των ανηλίκων, την θανατική ποινή. Ασχολούμεθα με την κατάσταση ασφαλείας στην νότιο-κινέζικη θάλασσα και επιθυμούμε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία πλαίσιο των περιφερειακών και των πολυμερών οργανισμών. Έχω λάβει πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Οι περισσότερες εξ αυτών ε, είναι θετικές και οι τροπολογίες αυτές εντάσσονται πολύ καλά στην ε, κατανομή της έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις εισηγήτριες για τις πολύ καλές προσθήκες και προτάσεις. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι και θα καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Υπάρχει μόνο μία τροπολογία όπου δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κανένα συμβασμό γιατί ε, τάσεται ε, κατά της συμφωνίας PCA. Και κατά τα άλλα θεωρώ ότι όσον αφορά τους συμβασμούς υπάρχει διαφορετική στάση ε, στην παράγραφο 6 ο μηχανισμός καταγγελιών ε, εκεί διαφωνούμε και στην παράγραφο 23 που αφορά στις ε, συγκρούσεις στη νοτιοκινέζικη θάλασσα. Αλλά όπως σας είπα στο βαθμό του δυνατού θα αναζητήσουμε το συμβιβασμό. Κατά τα άλλα επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι στην έκθεση εξακολουθούμε να θέλουμε την ε, νομική δεσμευτικότητα ανάμεσα στο PCA και τις ε, συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Υπάρχουν πολύ σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς εξακολουθούμε να απαιτούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών να την ελέγχει και κάτω από το πρίσμα της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς όπως το ζητάει και ο διαμεσολαβητής Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι είναι η τελευταία φορά του Trans-Pacific Agreement. Θα πρέπει λιγάκι να το δούμε και να ε, προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε μήπως ε, στην πρώτη συνεδρίαση των ε, σχεδόν εισηγητών μπορούμε να δεχτούμε κάποιες ε, τροπολογίες όσον αφορά αυτή τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ρηνικού. Αυτό που προηγουμένως αναφέρθηκε ως συμφωνία TPAC. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Λοχμπίλερ και τους σκιώδεις εισηγητές των υπολείπων πολιτικών ομάδων που εργάστηκαν επί της σημαντικής αυτής εκθέσεως. Η κύρωση της συνεργασίας ελληνικής σχέσης και συνεργασίας με ε, το Βιετνάμ είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους Βιετναμέζους εταίρους μας ε, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτήν την κύρωση. Πριν επικεντρωθώ σε κάποια από τα στοιχεία, θα ήθελα απλώς να ήθελα να ζητήσω από τους, από τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στον πειρασμό, να χρησιμοποιήσουν αυτή την έκθεση για να ε, επικρίνουν το Βιετνάμ ε, επί παντός επιστητού και σε κάθε λεπτομέρεια υπάρχουν ε, πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη για ε, το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας. Όμως εδώ μιλάμε για μια συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας που έχει βέβαια κάποιον αντίκτυπο γενικότερο στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε αυτές τις σχέσεις και να τις βελτιώσουμε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε το θέμα, για παράδειγμα, των δικαιωμάτων. Μπορούμε να το κάνουμε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ας μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Κάποια σημαντικά στοιχεία. Καταρχά, θα έλεγα είναι σημαντικό να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Το Βιετνάμ πρέπει να αναλάβει πολλές προκλήσεις για το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών. Το θέμα των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ειδικότερα στις ορεινές περιοχές, η αναθεώρηση του συστήματος της ε, ε, δικαιοσύνης και της ποινική δικαιοσύνη, γιατί αυτή τη στιγμή οι ε, ειρηνευτικέ δραστηριότητε ποινικοποιούνται λόγω για την εθνική ασφάλεια. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο πλαίσιο του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ ε, να ε, προσπαθήσουμε να βρούμε την πιο ρεαλιστική λύση για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε το Βιετνάμ σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ε, η συμφωνία ανταλλαγών, ε, ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών είναι πολύ σημαντική και για μας και για το Βιετνάμ, ειδικότερα για το θέμα της, για, για λόγους ανταγωνιστικότητας, επειδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν τώρα μια προνομιούχο πρόσβαση σε μια πολύ δυναμική αγορά Μιλάμε για 100 εκατομμύρια άτομα, μιλάμε για μια αγορά 100 εκατομμυρίων ατόμων ε, μιας τεράστιας, ε, ενός τεράστιου δημογραφικού δυναμικού. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν το Βιετνάμ να ε, ενισχύσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων εξαγωγών στην αγορά τη μέσω καταπολέμησης της διαφθοράς που είναι μια τεράστια μάστιγα σε αυτή τη χώρα όπως και σε άλλες χώρες βέβαια. Αυτό βέβαια θα ενθαρρύνει και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΖΕΑΝ ε, και νομίζω ότι είναι επίσης εποφελές και για τη διαφάνεια του οικονομικού τομέα και τη μακροοικονομική ε, συνεργασία μας. Το Βιετνάμ είναι σημαντικός εταίρος ε, στην περιφερειακή γεωπολιτική, ειδικότερα όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν ε, στην θάλασσα της Κίνας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. βέβαια, ο ρόλος μας δεν είναι να κατακρίνουμε, αλλά να βρούμε μια ειρηνική λύση μεταξύ όλων ε, μεταξύ όλων ε, των χωρών της διεθνούς κοινότητας. Ε, επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρξει ένας κώδικας διοντολογίας σε περιφερειακό επίπεδο και αυτή η συμφωνία είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας και τους, τις αρχές μας της ειρήνης, της θαλάσσιας ασφάλειας όπως επίσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να συνεχίσουμε τη ε, συνεργασία μας με τη συνάδελφο Λοχμπίλερ. Ε, την ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να μείνω στο τέλος συνεδρίασης γιατί έχω αργήσει δυστυχώς ε, σε άλλες επιτροπές που πρέπει να παραστώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ο κύριος Μπετίνη, για την εξαιρετική της δουλειά. Εγώ υποστηρίζω μεθαίνω στην κύρωση αυτής της συμφωνίας και συμφωνώ και με τον κύριο Πρέντα υπό την έννοια ότι το Βιετνάμ αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που κινείται πολύ, είναι μια χώρα την οποία είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ επανειλημμένος. Ε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε κοινωνικό επίπεδο, είναι πολύ ζωντανά και ανοιχτά τα πράγματα και πρέπει να δούμε και την κατάσταση να μεταρρυθμίσουμε, κυρίως όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ε, λάβουμε υπόψη μας και τις τραγωδίες που βίωσε η χώρα στο παρελθόν και παρά το γεγονός ότι ένα ουσιαστικό τμήμα του λαού του Βιετνάμ δεν τα θυμάται καν αυτά τα πράγματα γιατί το Βιετνάμ είναι μια νέα χώρα και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που γεννήθηκε μετά από το τέλος ε, του πολέμου με τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής, αλλά αυτό είναι ένα παρελθόν που ακόμα και τώρα, κυρίως ε, στη βόρεια πλευρά της χώρας, έχει σημαδέψει τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συμφωνία ώστε να προσπαθήσουμε να ανοίξει ακόμα περισσότερο η οικονομία της Βιετνά, του Βιετνάμ, η κοινωνία του Βιετνάμ και να δώσουμε μια όθηση προς ε, τις μεταρρυθμίσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα οποία έκανε η συνάδελφος είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θα σας ε, σχολιάσω αναλυτικά τις τροπολογίες που υπέβαλα. Ελπίζω κάποιες να συζητηθούν ε, ή να συμπεριληφθούν σε κάποιο συμβιβασμό και να ληφθούν υπόψη και πιστεύω ότι εμείς κάνουμε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική εταιρική πράξη προς τη σωστή κατεύθυνση κύριε Πρόεδρε. ο κύριο Τάνοκ, ε, εκ μέρου τη Ευρώπη των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ε, και του σκιώδης ηγητή που δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί ε, έχει κάποια άλλη υποχρέωση, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λοχπίρερ για την εξαιρετική της έκθεση. Έχουμε την 25η επέτειο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Με την πάροδο των ετών ήμουν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο Βιετνάμ, κυρίως ε, την δικτατορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την πραγματικότητα του Βιετνάμ, το Βιετνάμ τώρα συντονίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει στην ΑΣΕΑΝ και η ΑΣΕΑΝ είναι μια εμπορική ε, λέσχη και έχει ε, εταίρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και από πολιτικής και από οικονομικής κοπιάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως ε, λαμβάνεται και άμεση ενίσχυση και θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2020 Επομένως είναι πολύ στενή η δεσμή με το Βιετνάμ και η πολιτική μου ομάδα σίγουρα επικροτεί την υπογραφή αυτής της ε, συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε το γεγονός ότι παρά ε, τις ε, μεγάλες επιτυχίες που είχε το Βιετνάμ όσον αφορά την ε, φτώχεια, την κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση, την παιδεία και την υγεία. Υπάρχουν θέματα, ε, πνευματικά δικαιώματα, παιδική εργασία, πρόσβαση στην εκπαίδευση και για μένα είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της θρησκευτική ελευθερίας και για τους βουδιστές και για τους καθολικούς και για άλλες ε, θρησκευτικές ομάδες, ε, ε, κυρίως ανθρώπους οι οποίοι μετά από τον πόλεμο του Βιετνάμ αλλαξοπίστησαν, καθώς επίσης και όλα όσα έμειναν ως κατάλοιπα. Υπάρχουν για παράδειγμα φυτοφάρμακα τα οποία είναι ακόμα στην περιοχή λόγω του πονέμου του Βιετνάμ και αυτά είναι προβληματικά στοιχεία σε μια χώρα όπως το Βιετνάμ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν μέσω του εμπορίου και της βοήθειας να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην κυβέρνηση του Ανόη ώστε να βελτιώσει τα εσωτερικά της ζητήματα. Αυτό το καταπιεστικό καθεστώς λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθεί και θα προτιμούσαμε να υπάρχει ένα δημοκρατικό πολυκομματικό Βιετνάμ στο μέλλον. Το γεγονός όμως ότι περνάει ποιο μια ελεύθερη οικονομία, κάνει ένα ένιγμα προς τις ξένες επενδύσεις, είναι ένα θετικό βήμα και εμείς από πλευράς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διαφορθήκαμε ιδιαίτερα για την Κίνα, για το Βιετνάμ και τις γείτονές τους χώρες και θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να υπάρχει περισσότερη δημοκρατία, καλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα και βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Θα υποβάλουμε και εμείς κάποιες για την έκθεση αυτή, όσον αφορά την ελευθερία για τις θρησκευτικέ μειονότητες, δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία και ε, τα όσα κάνει η κυβέρνηση εκεί ε, από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Αν ε, δούμε την πρώτη εκδοχή ε, του ψηφίσματος, θα λέγαμε ότι ήταν ε, πολύ επικεντρωμένη στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρχαν όμως πολλές τροπολογίες, τις οποίες συνυπέγραψαν οι φιλελεύθεροι, Προσπαθήσαμε να επιμείνουμε και σε άλλα θέματα, όχι μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε μέσω αυτών των τροπολογιών να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξή. Αυτή η συμφωνία είναι μια ευκαιρία να ε, είναι πλέον σε ένα άλλο επίπεδο η σχέση μας και μας δίνει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα και στο Βιετνάμ να προσφέρει μεγαλύτερη ευημερία στους πολίτες της. Ε, το Κογκρέσο το Αμερικανικό έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις πλέον με το Βιετνάμ και αν θέλουμε και εμείς να έχουμε αντίκτυπο ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην ηθικολογούμε όλη την ώρα, πρέπει να έχουμε μια επικοδομητική και ρεαλιστική προσέγγιση και με τις εμπορικές συμφωνίες τις οποίες αυτή τη στιγμή συνάπτουμε με τον Βιετνάμ νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ευρύτερη συμφωνία με την ΑΖΕΑΝ και γι' αυτό ακριβώς η ομάδα μου θα υποστηρίξει τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Um, I want to thank Mr. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την έκθεσή της, επειδή ε, όλο και μεγαλύτερη είναι η σημασία των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ. Εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογίες εκ μέλους των σοσιαλδημοκρατών που αντιμετωπίζουν κατά τη γνώμη μας πολλά, πολλά ε, θέματα τα οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασίας με το Βιετνάμ. Πολύ σημαντική λοιπόν είναι η στρατηγική σημασία της, ε, του Βιετνάμ για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το Βιετνάμ ε, έχει ταχθεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συμμετείχε στην ενίσχυση των ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ και είναι συντονιστής για το διάλογο και το, τη συνεργασία, κάτι το οποίο φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα κατά το 2015. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν, το οποίο αναφέρεται είναι η ένταση ε, με την Κίνα σε σχέση με την Νότια Κινέζικη θάλασσα. Αν θέλουμε να είναι ε, σημαντικός ο ρόλος του Βιετνάμ ε, και ο δικός μας ρόλος στην περιοχή, η ύπατη εκπρόσωπος πρέπει να είναι δραστήρια στην παρακολούθηση της ε, διαδικασίας, όπως επίσης και την υποστήριξη μιας καλής λύσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Έχουμε υποβάλει λοιπόν πολλές τροπολογίες σε σχέση με την αντιμετώπιση σημαντικών ε, προβλημάτων και ανησυχιών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, χρειαζόμαστε νομοθεσία για την παιδική εργασία, για το λαθρεμπόριο ανθρώπων, όπως επίσης και το ευρύτερο λαθρεμπόριο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν στο Βιετνάμ, γι' αυτό εμείς προτείνουμε μια ειδική ομάδα εργασίας ή Επιτροπή, για το θέμα αυτό του της ε, νομοθεσίας που πρέπει να υπάρξει στο Βιετνάμ στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για την επίλυση του προβλήματος του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στα θύματα αυτής της κατάστασης ε, στο Βιετνάμ. Και γνωρίζω ότι κάποια ζητήματα δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό ε, σχέδιο έκθεσης, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως την εισηγήτρια, γιατί τα συμπεριέλαβε τροπολογίες. Πρέπει να κάνουμε μια ισχυρή έκκληση προς το Βιετνάμ, να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις σε σημαντικούς τομείς. Όμως το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενός εργατικού δυναμικού που αυξάνεται κατά πάνω από ένα εκατομμύριο Αν δείξει την πολιτική βούληση το Βιετνάμ να προχωρήσει για σημαντικά ζητήματα που αναφέρονται στην έκθεση όπως η φόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και την ε, δημιουργία μιας περιεκτικής κοινωνίας, τότε θα βρούμε την τεχνική υποστήριξη για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Με, ενώ αυξάνεται ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός σε 400 εκατομμύρια για το Βιετνάμ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει την ορατότητα των ενωσιακών δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας το Βιετνάμ για να εξασφαλίσουμε το στρατηγικό δυναμικό δυναμικό αυτών των πόρων. Εγώ με χαρά θα περιμένω τις περαιτέρω συζητήσεις για την έκθεση αυτή, αλλά και για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπαν οι σκιώδεις ηγητές, οι απόψεις που ακούστηκαν ε, εκφράζονται και στις τροπολογίες και γι' αυτό το λόγο δεν έχω να πω κάτι φοβερό, δεν άφησα και τίποτα το καινούριο. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτά που είπε η κυρία Βάουτμαν από τους ε, φιλελεύθερου και το είπαν τώρα και οι σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή στο πρώτο σχέδιο δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία και δυστυχώς ε, στο πρώτο σχέδιο αναγκάστηκα να κάνω πολλές τροπολογίες γιατί ήταν όλα πάρα πολύ περιορισμένα. Βλέποντας λοιπόν το πώς γίνεται η στάθμιση, διαπιστώνω ότι έχουμε τώρα τροπολογίες για τη χρηστή διακήρυξη, για την αντιμετώπιση διαφθοράς, για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, για την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν για όλα αυτά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι εστιαζόμαστε μόνο και ούτε θα εστιαστούμε μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας είπα και στην αρχή, κατά την άποψή μου πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες απόψεις ε, σχετικά με αυτό το μηχανισμό καταγγελιών έτσι ώστε να βρούμε ε, κάποιο μηχανισμό, να δούμε και τι θα γίνει με τις συγκρούσεις στη Νοτιοκινέζικη θάλασσα. Πάντως εγώ να σας πω ότι γενικά είμαι αισιόδοξη ότι θα βρούμε συμβασμό σε όλα. Και όσον αφορά στη συζήτηση επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στη γραμματεία και να πω ότι η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα είναι στις 16 Νοεμβρίου. Άρα 9-10 ε, Νοεμβρίου εκεί γύρω θα έχουμε κάποια συνεδρίες των συντονιστών ε, και νομίζω αυτό θα είναι σκόπιμο γιατί κάπου εκεί ε, ή λίγο μετά θα επισκεφτεί η αντιπροσωπεία με το Βιετνάμ επιτόπου τη χώρα, άρα θα ξέρουμε και τι ακριβώς έχει γίνει. η έκθεση τώρα για τις ε, Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες ε, είναι μια στρατηγικά και οικονομικά ε, ιδιαίτερα σημαντική χώρα. Γι' αυτό λοιπόν προτίθεμαι να σας προτείνω να αποφασίσουμε θετικά. Οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι οι Φιλιππίνες ε, λόγω της εσωτερικής της ε, δομής ε, μαστίζεται και από εσωτερικές έρηδες οι οποίες σχετίζονται με την αύξηση του Ισλαμισμού. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όσον αφορά στις Φιλιππίνες ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η ε, διαδικασία ειρήνης, ε, η εσωτερική διαδικασία ειρήνης. αυτήν πρέπει να τη στηρίξουμε τη διαδικασία, διότι οι Φιλιππίνες από το 2001 συμμετέχουν στη Διεθνή Συμμαχία κατά της ε, τρομοκρατίας. Άρα είναι μια χώρα πολύ σημαντική. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε και ότι η στρατηγική ανάπτυξη της ε, περιοχής σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα στη νοτιοκινέζικη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν η χώρα αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί σε σημαντικό μας εταίρο. Νομίζω ότι οι έρηδες όπως σας είπα που υφίστανται στην περιοχή θα πρέπει να διευθετηθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και να υπάρξει διεθνής διαμεσολάβηση. Οι Φιλιππίνες είναι το αντίβαρο του μεγάλου γείτονα και γι' αυτό είναι σημαντικό Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στη θάλασσα Μινανάου να είμαστε προσεκτικοί, να μην υπάρξουν αρνητικές ε, συνέπειες από αυτή τη συμφωνία που έχει συναυτεί. Οι Φιλιππίνες ε, έχουν πλέον μια ειδική προτιμησιακή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τη στηρίξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα χαρώ πάρα πολύ μετά τον καθορισμό της ε, καταληκτικής ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών ε, να συνεχίσουμε τη συζητήση μας για τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα να συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπετίνη. Εγώ την έκθεση αυτή κύριε Πρόεδρε τη ουσκό εξαιρετική και πολύ τολμηρή. Πιέζει τα πράγματα προς τα μπρος και συμφωνώ πολύ με αυτή τη στάση. Θα ήθελα να επισημάνω ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό να το επενθυμίσουμε στους αδέλφους. Οι Φιλιππίνες ε, τα τελευταία χρόνια έχουν ε, κάνει μια εκβάθρον αλλαγή. Ήταν μια χώρα πολύ ανασφαλής, ε, ε, που την είχε πλήξει διαφθορά, με πάρα πολλές συγκρούσεις, με ε, ε, περιοχές ε, εκτεταμένες κοινωνικής περιθωριοποίησης. Προς Θεού δεν εξαφανίστηκαν όλα τα προβλήματα διαμιάς, αλλά τα αποτελέσματα της Προεδρίας Ακίνο ήταν σημαντικά και έφεραν μια νέα προοπτική στη χώρα και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο πιο σταθερές και πολύ πιο αξιόπιστες. Επομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις Φιλιππίνες να τις προωθήσουμε με όλες τις χώρες αυτής της περιοχής της Ασίας. Οι Φιλιππίνες έχουν μεγάλο πληθυσμό, έχουν μια γεωπολιτική στρατηγική θέση πολύ σημαντική και πρέπει να πω ότι από αυτές τις χώρες ε, της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας ε, είναι η χώρα με την οποία έχει τις περισσότερους ιστορικούς δεσμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα απλώς να πω ότι βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τροπολογίες ε, βάσει της πείρας μου στις σχέσεις με τις Φιλιππίνες θεωρώ ότι θα πρέπει να πιέσουμε πολύ στο θέμα των πολιτιστικών ανταλλαγών. Ε, το συζητήσαμε και στην ΑΣΕΑΝ. Ε, στις Φιλιππίνες υπάρχει για παράδειγμα ε, ιστορικά πολύ καλός κινηματογράφος. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά διανομής και παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και η ΑΣΕΑΝ οργανώνεται σε κινηματογραφικό επίπεδο και σε άλλα πολιτιστικό γεγονότα ως μια ενιαία λεκάνη. Και νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι το οποίο υπάρχει ήδη, αλλά να το διευκρινίσουμε λίγο ακόμα καλύτερα και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. ES have asked them. They have nothing to say. Oh, they... Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάτι να πούνε. Ε, έχετε αλλά δεν θέλετε. να πω δύο λόγια για την έκθεση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι συμφωνίες είναι ένας τρόπος να αναβαθμίσουμε, να διευρύνουμε και να διαφοροποιήσουμε τις σχέσεις μας με διάφορες τρίτες χώρες και θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει γίνει πολύ καλή πρόοδος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Φιλιππινών σε αρκετά ζητήματα στο πρόσφατο παρελθόν. Ε, το Δεκέμβριο του 2014 υπήρξε μία ε, κίτρινη κάρτα η οποία ανακλήθηκε το 2015, η απαγόρευση του, ε, για την αλία ήρθε τον Ιούνιο του 2015 και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την υποστήριξη ε, που έδειξαν οι Φιλιππίνες στην φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Ασίας. Όσον αφορά την έκθεση, έχω ελάχιστες παρατηρήσεις, τις οποίες εν μέρει έχω διαβιβάσει στη γραμματεία. Κάποιες είναι απλώς καθεστώς γεγονότα, ε, ο αριθμός των Φιλιππινέζων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 800.000 και όχι 600.000. Στην παράγραφο 10 της έκθεσης, που νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράγραφος, αναφερόμαστε στις, ε, ε, ε συμφωνίες GSP, στο Γενικό Προτιμησιακό Καθεστώς. Νομίζω ότι εκεί το θέμα είναι περισσότερο θέμα εφαρμογής και όχι έλλειψη κύρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, κύριε Μπετίνη. Αυτά που μας είπατε θα τα λάβω ιδιαίτερα υπόψη μου και σας παρακαλώ να καταθέσετε τις σχετικές τροπολογίες για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να ολοκληρωθεί η έκθεση. Τώρα τι θα κάνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Hmm? But 20 Διάλειμμα 20 λεπτά για να πιείτε καφέ και να πιείτε κονιάκ, λέει ο πρόεδρος. The liberals, they have the most Αυτό βεβαίως αφορά τους ελεύθερους, γιατί αυτοί είναι οι πλούσιοι. Εμείς οι άλλοι δεν έχουμε. Κύριε Μπετίνη, πρόεδρε, συγγνώμη, Κάτι ξέχασα, ξέχασα να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως ε, στη συζήτηση για τις Φιλιππίνες ετέθηκε το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Εξακολουθεί να ισχύει, υπάρχει κάποιο άλλο, είναι τεχνικής φύσης η ερώτησή μου. Αυτή ήταν η συζήτηση και κανείς δεν ζήτησε το λόγο. Συγγνώμη πρόεδρε, άλλο δεν, δεν εννοούσα αυτά που απαντάτε. Συγγνώμη, αναφέρομαι στη σχέση και στην έκθεση για τις Φιλιππίνες. Εκεί υπήρχε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ξακολουθούν υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με τους Φιλιππινέζους ε, για το πρόγραμμα και θα σας το ανακοινώσουμε τις επόμενες εβδομάδες όταν ε, θα έχει γίνει συζήτηση και θα έχουμε δει λιγάκι τις ε, τροπολογίες πριν καταλήξουμε στα τελικά μας συμπεράσματα. Γύρω στο Νοέμβριο θα γίνει αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διακόπτεται η συνεδρίαση.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 και θα μας ενημερώσει κατά κύριο λόγο για την χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Και δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο. Ίσως ε, μπορούμε να συζητήσουμε και τη συνεργασία ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών που την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω Τετάρτη Πέμπτη ήτανε, κατέληξε σε κάποιες καλές εξελίξεις ε, για τα θέματα της ε, μετανάστευσης και της ε, διατομεακότητας, δηλαδή με την έννοια ότι πολλοί τομεί είναι αρμόδιοι πλέον και πολλές ε, υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τους μετανάστες. Ίσως μπορούμε να συζητήσουμε και για αυτά. Πάντως ε, να μην χάσουμε άλλο χρόνο και θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στην κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλμαρ. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που έχασα ε, την ολομέλεια του Κοινοβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Ε, ε, όμως συνήλθα, μου φαίνεται είχαν πέσει λίγο οι μπαταρίες στον οργανισμό μου. Πάντως τώρα είμαι καλά και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Εχθές είχαμε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πολλά σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, με αυτά, λέγοντας αυτά που πάει και χθε στους Υπουργούς Εξωτερικών με δύο σημεία τα οποία δεν ήταν τμήμα της ημερήσιας διάταξης, αλλά ε, είχαν αναφερθεί στις σύντομες ε, εισαγωγικές μου παρατηρήσεις εχθές. Το ένα είναι η προσοχή που δώσαμε στις εκλογές στη Λευκορωσία. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά κατά τις επόμενες εβδομάδες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε για τις κυρώσεις που ε, θα επιβληθούν και επίσης η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στην Ιερουσαλήμ, ε, τη Δυτική Όχθη, στη διόρυγα της Γάζας και αυξανόμενη ε, ένταση στην Μέση Ανατολή. Το είπα και στους Υπουργούς Εξωτερικών και σας το λέω και τώρα ότι ο ε, πρόεδρος Αμπάς και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου μου τηλεφώνησαν την Κυριακή το βράδυ για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την ένταση που έχει αυξηθεί ε, στην περιοχή, να προσπαθήσουμε αμέσως ε, να προχωρήσουμε στη διαδικασία την οποία συμφωνήσαμε ε, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ε, Γενικής ε, Συνέλευσης του ΟΗΕ, να υπάρξουν συγκεκριμένα βήματα επιτόπου συνεπή σε σχέση με τις συμφωνίες μας για να μπορέσουμε να δώσουμε έναν ορίζοντα ελπίδας και στους Παλαιστίνιους και στους ε, οι Ισραηλινούς να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση στην Ιερουσαλήμ που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και εκτός ελέγχου. Τέσσερα σημεία είχαμε στην ημερήσια διάταξη εχθές ε, που είχαν κατά κάποιο τρόπο σχέση το ένα με το άλλο. Ε, Λιβύη, Συρία, ε, κρίση μεταναστευτική και προσφυγική και επίσης οι ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ 20 χρόνια μετά με την εκπνοή της Συμφωνίας του Κοτονού ε, ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό της εξωτερικής δράσης και της εργασίας που έχει να κάνει με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με τις ριζικές αιτίες. Ε, η Συρία και η Λιβύη είναι οι δύο δύσκολες επίμαχες καταστάσεις στην γειτονιά μας από όπου προέρχονται οι ροές και βεβαίως το θέμα του προβληματισμού μετά από, τον κοτονού, μετά από το κοτονού έχει να κάνει και με προβληματισμό διαφόρων εταίρων σε όλο τον κόσμο, ε, με τους οποίους έχουμε συμφωνίες που μπορούν να επιτρέψουν ε, την ε, επιστροφή, την επανεισδοχή και όλα αυτά τα σημεία, εν πάση περιπτώσει που σας ανέφερα, συνδέονται μεταξύ τους. Θα αρχίσω με τη Λιβύη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αφορούν και τη Λιβύη και τη Συρία και το θέμα το προσφυγικό. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους υπουργούς, ε, να μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα σημαντικό ισχυρό μήνυμα καταρχάς προς όλους τους ε, πολίτες της Λιβύης, να τους ε, ζητήσουμε να εγκρίνουν τη συμφωνία που βρίσκεται επιτάπητος αυτή τη στιγμή. Επίσης ενημερώσαμε και το χρονοδιάγραμμά μας ε, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2015 για την ε, υποστήριξη με, όλες τις πιθανές, ε, με όλους τους πιθανούς τρόπους όταν θα αρχίσει να υπάρξει μια, μια κυβέρνηση εθνικής ομόνιας δεν ε, μπορώ να σας πω πάρα πολλέ λεπτομέρειε για τι ημερομηνίε, Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ είχα προτείνει στου υπουργού Εξωτερικών, όπως θα θυμάστε, ενδεχομένως να αρχίσουμε να δουλεύουμε το πακέτο υποστήριξη ενδεχομένη υποστήριξης ε, ε, στη Λιβύη το Φεβρουάριο. Ήμασταν έτοιμοι το Μάρτιο εγκρίναμε ένα ε, χρονοδιάγραμμα, ένα προγραμματισμό ήδη το Μάρτιο, σε περίπτωση που η κατάσταση στη Λιβύη μας ξεπερνούσε, αλλά δυστυχώς δεν ε, συνέβη αυτό, δεν μας ξεπέρασαν οι εξελίξεις. Είναι πάντως καλό να μπορούμε να ε, διαπιστώσουμε ότι ήταν αρκετά προχωρημένος ο προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν προκειμένου. Δεν ε, θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ε, καταρχάς, γιατί είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει από κοινού με τους εταίρους μας στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες εναλλακτικέ επιλογές σε, διάφορες, σε διάφορους πιθανούς τομείς. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους Δήμους, πώς να τους υποστηρίξουμε σε σχέση με τις κεντρικές υπηρεσίες. Μόλις το συζήτησα αυτό πριν από μερικούς, ε, πριν από μερικά λεπτά και συγγνώμη που καθυστέρησε κιόλα για να έρθω εδώ με την Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών το συζήτησα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητάω και μαζί σας, αλλά και με, τους, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, πώ μπορούμε επιτόπου να υποστηρίξουμε τους Δήμους και τις κοινότητες στη Λιβύη, όχι μόνο από απόψεω ασφάλειας, αλλά και παροχή υπηρεσιών. Αλλά θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε όλα αυτά με ε, τις αρχές της Λιβύης ε, όταν σύντομα ελπίζουμε ε, πρώτα ο Θεός, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό. Και να δούμε επίσης και πώς πάει το θέμα της επιχείρησής μας κατά της, ε, του λαθρεμπορίου ε, στην Μεσόγειο, την επιχείρηση Σοφία. αυτό ήταν το όνομα του παιδιού που γεννήθηκε πάνω σε ένα γερμανικό πλοίο που συμμετείχε στην επιχείρηση και αυτό το κάναμε για να δείξουμε ότι ενώ ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι προφανώς να καταπολεμήσουμε τους λαθρεμπόρους και τα εγκληματικά δίκτυα, ε, μια παρενέργεια η οποία είναι ένα καθήκον οποιοδήποτε επιχειρεί στη θάλασσα είναι να ε, σώζουμε χιλιάδες ε, ζωές και στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τα καταφέραμε και τα καταφέραμε μάλιστα μεταξύ των ε, διασωθέντων ήταν πολλά νεαρά παιδιά. Την Παρασκευή εγκρίναμε την επιχείρηση αυτή, την εντολή, το πεδίο εφαρμογής της, την πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο της φάσεις 2. Ε, αυτό το είχαμε κάνει πριν περάσει το ε, ψήφισμα. Ε, κατά τη γνώμη μου, από πολιτικής απόψεις, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, μήνυμα αυτό, το γεγονός ότι υπάρχει μια συνολική υποστήριξη για την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, για την καταπολέμηση αυτών των λαθρεμπόρων που διακινούν ανθρώπους. Και είναι επίσης ιδιαίτερο σημαντικό το γεγονός ότι όχι μόνο πέρασε το ψήφισμα, αλλά με 14 ψήφους υπέρ και μία μόνο αποχή πέρασε ε, αυτή της Βενεζουέλας και ελπίζω ότι αυτό μας ε, δίνει σε όλους τη δυνατότητα αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ε, προχωρήσουν και να ξεχάσουν αυτό το, την ιδέα που είχαν ότι η Κίνα και η Ρωσία ήταν κατά 14 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος ε, αποχής, ε, κάτι το οποίο δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να συνεργαστεί περαιτέρω για το πώς θα προχωρήσουμε. Προφανώς βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, με τον τρόπο ίσως που έχουμε συνεργαστεί κατά, τα τελευταί, κατά τους τελευταίους μήνες, ε, με τον τρόπο που έχουμε συζητήσει με τους συνομιλητές μας, τους τελευταίους μήνες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο στάδιο της φάσης 2 υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε και ελπίζω ότι η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό είναι επίσης και η υποστήριξη των αρχών της Λιβύης, ε, κάτι ε, το οποίο ισχύει, δηλαδή έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συνεργαστούν μαζί μας προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά όσον αφορά στη Λιβύη, όσον αφορά στη Συρία τώρα. Καταρχάς ε, υπήρχε ένα ευρωπαϊκό ε, ε, υπήρχε μια ευρωπαϊκή ε, ενότητα. Ε, εγώ προσωπικά δεν, ανησυχούσα, αλλά είναι σημαντικό να διαπιστώνει κανείς ότι όντως υπήρχε μια ενότητα. Την είχαμε διαπιστώσει ήδη πριν από την συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών. Είχαμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Επίσης είμαστε και πολύ ενωμένοι επί τριών πτυχών συνολική στρατηγική για τη Συρία και για την, το ρόλο της Ένωσης για τη συμμετοχή συμμετοχή της επίλυσης της ε, Συριακής ε, κρίσης, ε, ανθρωπιστική πτυχή, πτυχή ασφαλείας και πολιτική πτυχή. Από απόψεως ανθρωπιστικής ε, θα το γνωρίζετε όλοι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, και θα είμαι πολύ σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος δωρητής και αποφάσισε μάλιστα μόλις προσφάτως να αυξήσει κατά αξιόλογο ε, ποσοστό τη συμμετοχή της και προς τις υπηρεσίες του ΟΗΕ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και αναφέρομαι κυρίως στην ύπατη αρμοστία ε, αλλά και την ενίσχυση της υποστήριξης στις εθνικές και τοπικές αρχές ε, που φιλοξενούν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Αναφέροντας ε, αυτές τις αρχές, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι φιλοξενούνται όχι σε στρατόπεδα, αλλά σε τοπικές αρχές. Οπότε άμα θέλουμε να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες και να υποστηρίξουμε και ε, τις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν ε, αυτά, ε, αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε όχι μόνο υλικά αλλά και, και, και με υλικό τρόπο και στη Συρία και στο Λίβανο. Από ανθρωπιστικής απόψεως λοιπόν έχουμε αυξήσει την συμμετοχή μας ε, σε μεγάλο βαθμό. Ε, επίσης, ε, ξέρετε ότι υπάρχει και ένα ταμείο, είχα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να ενισχύσουν αυτόν τον προπολογισμό, κάτι το οποίο σιγά-σιγά συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου πολύ σιγά, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα φερθούν την πέμπτη περαιτέρω αποφάση στο Συμβούλιο ε, ως προς αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω για το ανθρωπιστικό κομμάτι ότι εξακολουθούμε να συνεργόμαστε, ε, με, να συνεργαζόμαστε ε, στο σύνορο μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, είναι δύσκολη η κατάσταση. Παρόλα αυτά υπάρχει ε, υπάρχει δυνατότητα συζήτησης με τις περιφερειακές αρχές εκεί για να μπορέσουμε να ζητήσουμε ανθρωπιστική πρόσβαση και σεβασμό του διεθνούς ε, ανθρωπιστικού δικαίου. Ελπίζουμε ότι, είναι πολύ σημα... ότι, είναι... ότι αυτό θα συμβεί γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική ε, εξέλιξη. Η μεγαλύτερη προσοχή της κοινή γνώμης αλλά και, της, ε, ε, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αφορά κυρίως τις ρωσικές κινήσεις. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο αυτή ε, τη στιγμή. Έχουμε σαφές δηλώσεις, σαφείς δηλώσεις στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που μπορεί ήδη να τα διαβάσετε. Ήδη δηλαδή από χθε αναφέρθηκε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι όλες οι στρατιωτικές παρεμβάσεις πρέπει καταρχάς ε, πρέπει να αφορούν την Αλνούσρα, ε, το Ισλαμικό κράτος και άλλους αναγνωρισμένους τρομοκρατικούς οργανισμούς, ε, τρομοκρατικές οργανώσεις και όχι με άλλους τρόπους, σε, άλλους, σε άλλες συνθέσεις αντίστασης ή ομάδων αντίστασης και λοιπά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πλήρως συντονισμένες μεταξύ των διαφόρων διεθνών και περιφερειακών εταίρων που παρεμβαίνουν ε, στρατιωτικά στην καταπολέμηση του ΝΤΑΕΣ ε, μερικές φορές αυτό ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει και έχουμε εκφράσει πολύ σοβαρές ανησυχίες, ε, ειδικότερα όσον αφορά την παραβίαση του εναερίου χώρου της Τουρκίας ε, που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη κλιμάκωση και πολύ σοβαρά ατυχήματα και είναι κάτι που το συζητήσαμε επίσης και με τον πρόεδρο Ερντογάν όταν ήρθε την περασμένη εβδομάδα εδώ στι Βρυξέλλες. Και τρίτον, ε, και πρέπει να ε, το γνωρίζουμε αυτό, τα συμπεράσματα χθε το ε, ανέφεραν σαφέστατα. Δεν υπάρχει κανένα, καμία ε, περίπτωση ε, στρατιωτική δράση στην οποία δεν συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ, ε, με πάση ούτε πρόκειται να το κάνει στο άμεσα προβλέψιμο μέλλον, ε, ακόμη και αν συμφωνεί και συμμετέχει στην προσπάθεια κατά του Νταές, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αποδυναμώσουμε τις ελεύθερες περιοχές, ειδικότερα στο Ιράκ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η στρατιωτική δράση κατά του ΝΤΑΕΣ να, ε, να προκαλέσουν το τέλος της κρίσης από μόνες τους. Συμφωνήσαμε σε αυτό και επικεντρωθήκαμε χθε με τους Υπουργούς Εξωτερικών στον δικό μας ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργοποιήσουμε την ε, πολιτική διαδικασία της δημοκρατικής μετάβασης που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου και μάλιστα αναφέραμε στα συμπεράσματα, υποθέτω λάβατε γνώση, την ανάγκη ενεργά εκ των προτέρων ε, ε, με πολύ αποφασιστικό τρόπο να συμμετέχουμε ε, από κοινού με τον ΟΗΕ στη διαδικασία του ΟΗΕ. Δεν εννοούμε ότι κάποιος άλλος πρέπει να κάνει τη δουλειά για μας. Ε, αντιθέτως, η δική μου ταπεινή ε, εμπειρία Δύο μπορεί να είναι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς, την, προς τον ΟΗΕ απόσταση. Μπορεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ, την υποστηρίζουμε, ε, την εξετάζουμε, αλλά μπορούμε και να ε, εμπλακούμε, γιατί ξέρετε, ότι του ΟΗΕ είναι τόσο ισχυρή όσο τους κάνει η διεθνή, σκηνή, η διεθνής γνώμη. Και χθε αυτό που αποφασίσαμε είναι μια ουσιαστική συμμετοχή, εμπλοκή από πλευρά μας και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι να συμμετέχω και να ενισχύσω την ε, προσπάθεια του ειδικού αποσταλμένου για τη Συρία ε, να προσπαθήσει να επηρεάσει τις περιφερειακές αρχές να τις υποστηρίξει και να αρχίσει η πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη, μετάφαση, στη μετάβαση. Ε, άρχισα να το κάνω αυτό μόλις σήμερα το πρωί όταν, ε, όταν ε, ε, υποδέχθηκα μία αντιπροσωπή από το Ιράν, αρχίσαμε να το συζητάμε, συζητήσαμε πάρα πολλή ώρα, είχαμε νεανότερους αξιωματούχους συζητήσεις και από τις δύο πλευρές ε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ε, ε, πολιτική αυτή διαδικασία και είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε με όλους τους εταίρους, Ιράν, Σαουδική Αραβία, τις υπόλοιπες χώρες του Περσικού κόλπου, την Τουρκία ε, σε διεθνές επίπεδο, Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλου, όλα τα μέσα που έχουμε, διπλωματικά και πολιτικά, για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τους ε, εταίρους της Συρίας και τις, τα εμπλεκόμενα μέρη στη Συρία ώστε να μπορέσει να αρχίσει η πολιτική διαδικασία. Ως προς τη μετανάστευση τώρα, που ήταν το τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας, είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σε ένα μόνο έγγραφο προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε εδώ και πολλούς μήνες, ε, ε, ό,τι κάναμε εμείς για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων, προσπαθήσαμε να ε, δούμε τις δύο διαδρομές, την νότια και την ανατολική, Εκεί επικεντρώσαμε την προσοχή μας και προσπαθήσαμε να ε, λάβουμε και υπόψη ε, τα απορίσματα της ε, διάσκεψης υψηλού επίπεδου για την Ανατολική Μεσόγειο που συνήλθε και την περασμένη εβδομάδα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ε, εταίρους μας ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι δύσκολη η δουλειά μας ε, και η συνεργασία μας με την Τουρκία για το θέμα αυτό και αυτό έχει άμεση σχέση με τη συζήτηση που είχαμε για τη Συρία. Πρέπει επίσης να επιστρατεύσουμε όχι μόνο την οικονομική υποστήριξη αλλά να αυξήσουμε και τη χρήση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των χερσαίων συνόρων και ε, την ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και μεγαλύτερη συνεργασία με τις υπηρεσίες ε, του ΟΗΕ, για παράδειγμα την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, επειδή οι ροές από τη Συρία αφορά κυρίως πρόσφυγες και τούντες άσυλο έχουμε επιμείνει πάρα πολύ στην ανάγκη αύξησης ε, και προσπάθειας ε, ύπαρξης επιχειρήσεων ε, προς όφελος της αστυνομικής συνεργασίας, ειδικότερα για την καταπολέμηση των λαθρεμπόρων, γιατί αυτό είναι κάτι που στην νότια διαδρομή μέσω της Μεσογείου έχουμε αντιμετωπίσει με αρκετά αποφασιστικό τρόπο κατά τους τελευταίους μήνες μέσω των θαλάσσιων επιχειρήσεών μας και με τους βασικούς μας εταίρους ε, ειδικότερα στην υποσαχάρια Αφρική, αλλά προς, στην ανατολική διαδρομή έχουμε πολύ ακόμη δουλειά για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ε, διακινητές, τους λαθρεμπόρους ε, της ανατολικής διαδρομής. Όσον αφορά τώρα ε, την προετοιμασία της ε, Συνόδου της Μάλτας, προσπαθούμε όχι μόνο να προχωρήσουμε με το θέμα του νέου ταμείου, αλλά να δούμε και τι ακριβώς πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτό το ταμείο, ποια ακριβώς προγράμματα, ώστε να είναι καλύτερη η εφαρμογή τους και σαφέστατη. Είπα μάλιστα και στους υπουργού Εξωτερικών εχθές ε, ότι υπάρχουν τρόποι να συνεργαστούμε περισσότερο με τη συμμετοχή των κρατών μελών για το διάλογο υψηλού επίπεδου που έχουμε αρχίσει κατά τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες με μια σειρά χωρών, κυρίως της Βορείου Αφρικής και της Υποσαχάριας Αφρικής. Ε, ε, θα πάω στην Αντίσα Μπέμπα την επόμενη εβδομάδα και έχω και κάποιους άλλους, ε, κάποιες άλλες επισκέψεις για διάλογο υψηλού επίπεδου πριν από τη σύνοδο της Βαλέτας. Όλα αυτά, Συρία, Λιβύη και συμπεράσματα που αφορούν τη μετανάστευση είναι τμήμα της διαδικασίας ε, ε, προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα έχει ακριβώ την ίδια μερίσια διάταξη την Πέμπτη. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί περισσότερο στο εσωτερικό κομμάτι ε, της δουλειάς ε, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ε, βασιζόμενοι στην, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών, αλλά εν πάση περιπτώσει τα συμπεράσματα για, τα χθεσινά για αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ε, αντανακλούν μια πάρα πολύ συλλογική προσέγγιση των Υπουργών Εξωτερικών μας. Και τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, ένα σημείο είχαμε στην ημερήσια διάταξή μας όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού εν ώψη των συμφωνιών μετά από τη Συμφωνία του Κοτονού έχουμε αρχίσει να ε, τις επεξεργαζόμαστε. Είναι ένα ε, κατά παράδοση θέμα των Υπουργών Ανάπτυξης. Θα το συζητήσουμε στις 26 Οκτωβρίου όμως ε, ζήτησα από τους υπουργούς να μην τα αφήσουν μόνο στους υπουργούς ανάπτυξης γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στη συνεργασία μας ε, με τις χώρες αυτές ε, από απόψε πρέπει να περάσουμε σε μια πολιτική εταιρική σχέση και όχι σε μια αυστηρά αναπτυξιακή σχέση. γιατί έχουμε τόσο πολλά κοινά ε, σημεία ε, και πολλά ε, συμφέροντα για τη μετανάστευση, για την ασφάλεια, για την αντιτρομοκρατία, για τις οικονομικές σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να περάσουμε από την πτυχή, την καθαρά αναπτυξιακή, να περάσουμε σε μια ε, πολιτική ε, διαδικασία έχει αρχίσει η διαβούλευση, είμαστε ακόμα στην αρχή, θα το συζητήσουμε, το συζητήσετε και εσείς εδώ φαντάζομαι, αλλά θα ήθελα να πω ότι τόνισα στους Υπουργούς Εξωτερικών ότι δεν αφορά μόνο το θέμα των ε, εταίρων τους από τα Υπουργεία Ανάπτυξη, αλλά και για εκείνους. Σταματώ εδώ, θα, με χαρά θα ακούσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον καθένα για ένα λεπτό, συμφωνείτε γι' αυτό, εκτός μικροφώνου κάποιο σχόλιο. Διαφωνεί ο κύριος Μπροκ. Η κυρία Καλνιέτα έχει το λόγο για ένα λεπτό και μετά ο κύριος Τάνο καλά θα κάνει να μιλήσει και αυτός για ένα λεπτό για να έχουμε χρόνο στη συνέχεια να μιλήσουν όλοι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διαδραματίσει ένα παγκόσμιο ρόλο, όχι από οικονομικής ε, σκοπιάς και από πλευράς ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και ως πολιτική ισχύς. Ε, και αν διαβάσω τα νέα τα οποία έχουμε από τη Συρία, βλέπω τη Ρωσία, τις Ηνωμένε Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, προβάλλεται, δεν φαίνεται. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για τη δική μας ευρύτερη γειτονία και η ελπίδα μου είναι εάν μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα πιο ενεργό ρόλο για την προώθηση μιας πολιτικής λύσης ε, Δέχομαι μεν ότι εμείς είμαστε ήπια δύναμη, δεν είμαστε στρατιωτική δύναμη, αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Μετά από την παρέμβαση της Ρωσίας η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκη και μόλις τώρα χρησιμοποιήθηκαν 50 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική λύση όταν διαπιστώνετε ότι ε, μάλλον πρόκειται για αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουιτ. Χαίρομαι που αναρώσατε κύριε Πρόσωπη. σα συγχαίρω για τα όσα κάνατε για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Η κλιμάκωση της βίας είναι πάρα πολύ ανησυχητική και για ε, το θέμα της πρόσβασης στους ιερούς τόπους είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ελοχεύει ο κίνδυνος να χειροτερέψουν πολύ περισσότερα τα πράγματα τις επόμενες ημέρες και καλό είναι να υπαχρεπνείτε επί του ζητήματος. Δεύτερον, όσον αφορά τους βερβαδισμούς στην Τουρκία, δεν ε, προλάβατε να αναφερθείτε σε αυτή τη φρικτή αποτρόπια πράξη, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να επανέλθει η ειρηνευτική διαδικασία στο κουρδικό ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε την έκθεση για το αεροσκάφος, για το MH17, η οποία θα εκδοθεί σε μερικές ώρες. Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο ε, το θέμα αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι απαντήσεις, αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα. Και επίσης για το Ιράν σίγουρα πρέπει να γίνει και μια διαζώση συζήτηση και όχι μόνο δημοσίωσης, αλλά οι περισσότεροι αναρωτιούνται τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να συμμετέχει το Ιράν μαζί μα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, τι μπορείτε να κάνετε εσεί ώστε να έχουμε κάποια απάντηση. Να το συζητήσουμε και διμερώς αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αύριο υπάρχει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση στην Ουκρανία και για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μίνσκ 2. Από πλευράς ε, Ουκρανικής ε, η Ρωσία δεν έχει κάνει τίποτα για τη συμφωνία με την έννοια ότι έχει μόνο αναβάλει τις τοπικές εκλογές ε, δεν έχει επαναφέρει τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ουκρανίας Υπάρχει εντωμεταξύ και η παρέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία. Ο ε, Ασάντ ε, πλέον έχει αποκτήσει περισσότερο βάρος για την αντιμετώπιση της Συριακής κατάστασης, κυρίως απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεταναστευτικές ροές. Θέλω λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε ότι ο διάλογος ε, με τον Πούτιν και τη Συρία και το θέμα της Ουκρανίας και Κρυμαίας δεν σχετίζονται. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα μεταξύ τους. Άκουσα μεγάλη χαρά ότι οι Ρώσοι πλέον δεν απειλούν να καταθέσουν ε, βέτο για επιχείρηση επιχειρήσεις ε, που θα λάβουν χώρα στη Λιβύη, στα ύδατα της Λιβύης για να αντιμετωπιστούν οι διακινητές. Όμως ε, πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία για να ε, εφαρμόσουν αυτές τις συμφωνίες επαναπροώθησης με την Ελλάδα και να παρεμποδίζουν τις μεταναστευτικές ροές στην ΚΟ μεταξύ άλλων και σε άλλα ελληνικά νησιά. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, η δική μου ερώτηση αφορά τις εκλογές ε, στη Λευκορωσία της Κυριακής. Ε, το ε, Συμβούλιο Υπουργών, κάποιοι υπουργοί ακούστηκαν θετικοί και αισιόδοξοι όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, ζητούν να αρθούν οι κυρώσεις έναντι της Λευκορωσίας. Αλλά όμως 30 αντιφρονούντες από χιλιάδες ε, εκείνων που παρατήρησαν τις εκλογές ίσως είναι πιο αξιόπιστοι. Ο πρόεδρος Λουκασένκο ουσιαστικά επαναπιβεβαιώθηκε στο θρόνο του για άλλα πέντε χρόνια και νομίζω ότι θα συνεχίσει και άλλα 24 χρόνια γιατί ο γιος του είναι 11 χρονών και με βάση την ε, ε, νομοθεσία της χώρας μπορεί κανείς να είναι πρόεδρος για 35 χρόνια. Άρα δηλαδή εξή κατάσταση. Ε, δεν μπορούσαν να ελέγξουν σε εκλογικούς καταλόγους. Ε, υπήρχε κακή διαχείριση του όλου συστήματος το να ε, ψηφίζει κανείς και να μετρέται αυτό σε διαφορετικά, από ό,τι κατάλαβα αυτό που ελέγχθη τη Δευτέρα να αρθούν οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ βεβαιασμένο και πολύ επιπόλαιο. Μήπως θα έπρεπε να συνδεθεί με κάποιες προϋποθέσεις και να υπάρχει μια αντελεχέστερη αξιολόγηση της κατάστασης που δεν είναι ούτε και τόσο δημοκρατική ούτε και τόσο διαφανής. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Thank you. Ε, μου είναι λίγο δύσκολο να πω ότι η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε ουσιαστικότερη παρέμβαση εισαγωγικά του ουσιαστικότερη στη Συρία με κάνει να φοβούμε στην περίπτωση που είχε στρατών και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι θα πηγαίναμε και εμείς. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχει μια δύναμη στην πολιτική της θα πρέπει να είναι η ηθική στην πολιτική της. Και αυτό έρχεται να δέσει και με το τι τρέχει στην Ιερουσαλήμ στην οποία αναφερθήκατε. Πότε είπαμε εμείς τους, ε, στους Ισραηλίτες τι στο καλό κάνουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έχουν, έχουν ουσιαστικά εξαλείψει κάθε πιθανότητα επιβίωσης του αραβικού πληθυσμού σε αυτή την περιοχή πολύ περισσότερο να είναι κάποτε η πρωτεύουσα της, ε, του, μελλοντικού κράτους των, των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ. Thank you and also thank you, Madam ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Υπατή, εκπρόσωπη κυρία Λοχμπίλερ. Η ερώτησή μου αφορά την Λιβύη. Είχα την χαρά να μεταβώ στη Τινησία την ε, ε, περασμένη εβδομάδα και μίλησα με ε, φιλάρχους από τη Λιβύη και μας είπαν όλοι ότι χρειάζεται μια συμφωνία και υπήρχε ένας μεγάλος κατάλογος με αντιρρήσεις όμως. Ε, υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος μιας από τις πιο ε, σημαντικές φυλές ε, με ιδιαίτερη επιρροή και από ένα σημαντικό πολιτικό κόμμα και δεν τους διαβουλεύτηκε κανείς. Ε, οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα είπαν ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται έρευνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ερευνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συνεχίσει μέχρι το 2016. Θα υποστηρίξετε αυτή τη συνέχεια. Επίσης, όταν ε, αναφερθήκαμε στην ε, αποστολή της EUNAFOR, πολλοί συμφώνησαν ότι δεν πρόκειται για αποτελεσματική λύση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το μοντέλο αυτών των λαθρεμπόρων και υπάρχουν κάποιες ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις διάσωσης ε, που μίλησαν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία και είπαν ότι ε, δεν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που διασώθηκαν μετά από την έναρξη αυτής της επιχείρησης. Πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή τη στρατιωτική προσέγγιση για την καταπολέμηση των διακινητών ενώ θα έπρεπε να ληφθούν άλλα μέτρα που θα αποδυναμώσουν τα όσα κάνουν οι διακινητές. Τώρα, στην περιοχή του Σαχέλ και του Νίγηρα, είπατε ότι χρειάζεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα πολλαπλών σκοπών. Θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το κέντρο πολλαπλών σκοπών, αυτό το multi-purpose center που αναφέρεται εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την είπατε εκπρόσωπο. Πρώτη ερώτηση για τη Λιφία. Η Ιουναφόρ ε, έχει κάποια ε, προγραμματισμό για επίγες ε, αποστολές και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση αν προβλέπετε και χερσαία επιχείρηση το συζήτησαν ούτως ή άλλως οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθών, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Επίσης θα ήθελα να ξέρω και τι γίνεται επί τόπου. Η λύση ε, στη Συρία δεν είναι ο Ασάντ, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία στην οποία να καλύπτεται και η πλευρά του Ασάντ, τουλάχιστον ε, επειδή του υπερασπίζονται και η Ρωσία και το Ιράν. Έχουμε λάβει γνώση κατάστασης. Ε, εμείς ε, τι μέτρα σκοπεύουμε να λάβουμε για να σταματήσει αυτή η στασιμότητα. Επίσης και τι πιέσεις ασκούνται ενώπιον των χωρών συνεργασίας του κόλπου, οι οποίες χώρες δεν έχουν διαδραματίσει τον συνεπή ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσουν και ως προς τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, διότι νομίζω ότι έχουν και πολιτιστικές ρίζες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην περιοχή. Τέλος, όσον αφορά τα εγκληματικά δίκτυα στα Βαλκάνια, σκοπεύετε να ενισχύσετε τις παρούσες αποστολές, αν μπορείτε να βοηθήσετε για να υποστηρίξουμε τις χώρες εταίρους μας επιτόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε για το θέμα της ε, Συρίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε θα συνεχίσουμε δηλαδή τη στρατηγική του Ομπάμα που είναι ο μόνιμος ε, πόλεμος που δεν οδηγεί πουθενά ποτέ σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή μήπως ε, υπάρχει μια τοπική σημαντική δύναμη η οποία συνεχίζει ένα πόλεμο που σε τελική ανάλυση ίσως έχει κάποιο αποτέλεσμα κατά του ISIS. Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα εξετάσει, να τα σκεφτεί, να συνεχίσει το διάλογο που είναι χρήσιμος, διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους γιατί ο ISIS πρέπει να ιτηθεί, είναι ο εχθρός της Ευρώπης. Κατόπιν, για τη Λιβύη. Θα ήθελα να γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα τι κάνουμε για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε οι εμπλεκόμενοι να συμφωνήσουν, ε, να υπάρχει ε, κάποια βούληση για να τελεσφορήσει η όλη προσπάθεια. Είμαι όμως απεσιόδοξος. Και κάτι άλλο τι προτιθέμεθα να κάνουμε συγκεκριμένα για να αναπτύξουμε δραστηριότητες και να διαλυθεί το διέξοδο. Τέλος, η ύπατη εκπρόσωπος ε, πολύ σωστά λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη, ρεκόρ γίνεται στη βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Αλλά σε τελική ανάλυση γιατί δεν υπάρχουν άλλοι που να καλούνται να βοηθήσουν πρώτοι κυρίως οι ομόθρησκοί τους γιατί δεν καλούνται να βοηθήσουν πρώτοι ε, αυτούς που φεύγουν από τις αιστείες τους. Ευχαριστώ πολύ. Η σταθερότητα της συμφωνίας με τη Λιβύη εξαρτάται και από τη συμπεριφορά των ε, εξουσίων. Και ερωτώ, όσον αφορά Τουρκία, Κατάρ, Τρίπολη, Σοδική Αραβία, Αίγυπτο σε σχέση με τον Μπρουκ, υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις. Στην περίπτωση λοιπόν που τηρηθεί η συμφωνία, οι δικές μας οι προσπάθειες πώς ακριβώς εξολογείται για να ξεφορτωθούμε την Αλκάιντα και τον Άισις ε, μέσα στη Λιβύη. Η Τρίπολη και το, το Μπρουκ ε, θα πρέπει ίσως ε, ε, να συγκρατήσουν τους Λίβιους ή μήπως θα πρέπει να ε, προσφέρουμε την υποστήριξή μας επί τόπου. Τι είδους προοπτικές υπάρχουν όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, Είπαμε ότι πρέπει να είναι περισσότερο παρούς η Ευρώπη σε αυτές τις εξελίξεις και όποιος το λέει θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεπής γραμμή των κρατών σχετικά με τις επιλογές. Αυτά σε σχέση με τον Ασάντ, με τη Λευκορωσία, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία. Έχω τώρα δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εγώ επισκέφθηκα πριν από λίγες μόνο ημέρες το Λίβανο και την Ιορδανία. Και εκεί εντόπισα δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι μοιάζει να υπάρχει αλλαγή προσανατολισμού από πλευράς προσφύγων. Δεν βλέπουν ε, να υπάρχουν ε, λύσεις, άρα δηλαδή ε, θα τεθεί ένα θέμα μαζικής μετανάστευσης. Κατόπιν, η κρίση της κυβέρνησης στο Λίβανο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και τα κονδύλια που εκταμιεύσαμε αυτά πώς θα χρησιμοποιηθούν από μια ανύπαρκτη κυβέρνηση. Και τέλος όσον αφορά τη Λιβύη καλά κάνουμε και ζητάμε την ε, ανάληψη ευθυνών ελπίζω να υπάρχουν θετικέ απαντήσεις και διερωτώ αυτό το σχέδιο της ε, συμφωνίας ε, δεν θα μπορούσε να έχει μια νομική βάση για να εκδοθεί ένα σχετικό ψήφισμα από πλευρά Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Φωτίγα, τρία πράγματα. Η Ουκρανία. Το γεγονός ότι δεν συζητάτε το θέμα αυτό στις συζητήσεις του Συμβουλίου με ανησυχεί. Δεύτερον, η Λευκορωσία. Σε σχέση με χθες, ε, ήδη είχαμε μία ε, δήλωση του ωσά για την έλλειψη δημοκρατικής διεξαγωγής των εκλογών και επίσης να σας πω ότι η Ρωσική Ομοσπονδία στις 30 ε, Σεπτεμβρίου επέβαλε επιπλέον κυρώσεις ε, για την Τελωνιακή Ένωση ε, και εκεί συμπεριέλαβανε και τη Λευκορωσία και την Αλληλεία από πλευράς Πολωνίας. Γιατί η UNAFOR ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται η επιχείρηση αυτή δεν είναι σαφές το πεδίο εφαρμογής του δεύτερου ψηφίσματος. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, το, η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί και ε, καλύπτεται στο ε, πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το δεύτερο αυτό ψήφισμα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει στη δεύτερη φάση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Εγώ είχα ακούσει και είχα διαβάσει, τον έφερε και κάποιο άλλο συνάδελφο και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε ότι και εσεί θα θέλατε να συγκαλέσετε μια διάσκεψη ε, για να προσφέρετε ένα κάποιο ρόλο διαμεσολάβηση. Θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερα πράγματα λοιπόν για το κατά πόσον ισχύει αυτό ε, για τη Συρία και για το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα η Ρωσία, η Σαϊδική Αραβία και το Ιράν να συζητήσουν επί του ζητήματο. Όσον αφορά την επίθεση στην Τουρκία το περασμένο Σάββατο. Έχω την εντύπωση ότι η βία την οποία παρακίνησε και το ίδια η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες ε, εν ώψη των εκλογών την 1η ε, Νοεμβρίου, κυρίως ε, κατά των γραφείων του HDP, του Φουλικουρδικού Κόμματος. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν επεκρίθηκε η όλη αυτή η διαδικασία. Διάβασε ότι εσείς ε, έχετε μία ε, όλο ένα και πιο στενή σχέση με τις τουρκικές αρχές, ότι είναι πιο στενή από ποτέ. Μήπως θα πρέπει να το επικρίνουμε το γεγονός αυτό και το γεγονός ότι υποκίνησαν τις επιθέσεις, ε, ε, ε ιδίως και ενώπισαν εκλογών. Και εγώ ε, εδώ είμαι. Θα ήθελα να ρωτήσω τη σχέση μας με τη Ρουσία και το ρόλο που παίζει στη Συρία. Είπατε ότι η Ρωσία επεμβαίνει, αυτό το σημειώνουμε. Η Ρωσία μόλις άρχισε να βομβαρδίζει στόχους που δεν ήταν του ISIS, είπαν ότι υπάρχει κάποιο στρατιωτικό στοιχείο και προχτές είπατε ότι ο ρόλος της Ρωσίας στη Συρία δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός. Ίσως υπάρχει μια παρεξήγηση, να εδώ τώρα έχει την ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσατε. Νομίζω όμως ότι είναι σωστό να καταδικάσουμε το βομβαρδισμό πολιτών και να αντιλητεύσουμε το γεγονός ότι η Ρωσία χτυπάει και άλλους στόχους και όχι στόχους του ISIS. Ελπίζω να το κάνετε αυτό εδώ σήμερα. Ο κύριος Μιλανμόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη και σας ευχαριστώ και για τα όσα μας είπατε. Όσον αφορά ε, το σχέδιο για την ε, αποστολή αυτή. Νομίζω ότι είχε και ένα δεύτερο τμήμα ε, και νομίζω ότι με την κλιμάκωση των επιθώσεων της Ρωσίας είναι δύσκολο να λάβετε υπόψη αυτή τη δεύτερη ε, φάση. με την κλιμάκωση λοιπόν των επιθώσεων της Ρωσίας θα ήταν λίγο δύσκολο να έχουμε τον Ασάντ να συμφωνήσει σε κάτι. Ε, εσείς μας είπατε ότι η θέση της Λιβύης τίνει να είναι κατακερματισμένη. κατακαιρματισμένη. Πώς βλέπετε τη θέση της μετριοπαθούς Συρίας εδώ. Ε, μακάρι να υπήρχε κάποια θετική στάση και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον εξετάζεται και αυτό το περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας ε, όσον αφορά τις επαφές ε, Παλαιστίνης-Ισραήλ, αν είχατε κάποιες ε, καλύτερες επαφές, αν είστε πιο απεσιόδοξοι, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για τις επαφές με τη Ρωσία και το τι μπορεί να γίνει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τη Λιβύη, κυρία Πατή, σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω πέραν από την ασφάλεια των Συρώνων για να δούμε τι γίνεται ε, με την συμφωνία και αν η συμφωνία δεν τηρηθεί. Ε, πότε θα δούμε τι γίνεται με αυτό το πόλεμο πληροξουσίων που ε, έχει σχέση και με το Ισλαμικό κράτος και τις άλλες τρομοκρατικές ομάδες και αφορά την ασφαλειά μας για τη Συρία και το Ιράκ. Μα είπατε ότι τα κράτη-μέλη, ε, τα δικά μας, δεν κάνουν στρατιωτικέ παρεμβάσεις. Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο στο Ιράκ προσφάτω. Παρεμβαίνουν, δεν συντονίζονται, ιδίω όσον αφορά στην προμήθεια στους πεσμεργά, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να τους προμηθεύουμε εξοπλισμό, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να συντονιστούν και να επιτρέψουν να του συντονίσετε εσεί στην πραγματικότητα δεν συντονίζονται ώστε καν να διασφαλίσουν ότι υπάρχει για παράδειγμα σχολείο στους καταβλισμούς προσφύγων, γι' αυτό ακριβώς και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ και φεύγουν από εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα και επίσης ε, να υποστηρίξουμε και ε, τα ρεύματα των προσφύγων. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το Συμβούλιο πώς ακριβώς αισθάνεται που ανακοινώθηκε ε, δημοψήφισμα για την Ρεπούμπλικα Σπέρσκα, Σέψκα που πρόκειται να λάβει χώρα πολύ σύντομα και επίση, αν πραγματικά ε, διεξαχθεί δημοψήφισμα, εσείς τι λέτε από αυτού. Να σας υπενθυμίσω ότι στη Βοσνία Ερτσεγοβίνη υπάρχει μια συμφωνία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό εντάσσεται στη διαδικασία σταθεροποίησης και εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος στο να υπάρχει ε, ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετακίνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση η οποία όμως κατά κάποιο τρόπο θέτει σε κίνδυνο τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πρόεδρος, ε, ε, λυπάμαι, αυτό δεν έχει σχέση με την τελευταία ε, συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών, άσχετο αυτό που ρωτήσετε. Ο κύριος Πλάνκοβιτς, κυρία Μογκερίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Σχετικά με τη μετανάστευση, ε, θέλω να πω το εξή. Ε, χτες ε, ήταν το Συμβούλιο και οι συνάδελφοί σας, Τίμερμανς και Χάν, θα μεταβούν επιτόπου στην Άγκυρα για να δουν τι γίνεται με το πρόγραμμα δράσης με την Τουρκία. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε το πώς μπορεί να λυθεί η μεταναστευτική κρίση στο ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων με την Τουρκία και ποια είναι τα αιτήματα των Τούρκων. Αυτοί τι θέλουν για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, για το να ανοίξουν περισσότερα κεφάλαια. Αυτό το να ε, διατηρηθούν επίσης οι μεταναστευτικές ροές όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές αιστείες της κρίσης, δηλαδή κοντά στη Συρία. Τι γίνεται με όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι λόγω της ε, Τουρκίας έχει καθυστερήσει η έκθεση πρόοδου, αναβλήθηκε από αυτή την εβδομάδα ε, σε κάποια άλλη. Κύριος Φρόντι, κυρία Μογκερίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως για αυτά που μας είπατε ότι δηλαδή τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στην ε, πολιτική διαδικασία στο γίγνεσθε στη ε, Συρία. Αυτό δεν έχει γίνει ε, μέχρι τώρα όσο είσαστε στην εξουσία. Ένα από τα προβλήματα της περιοχής είναι ότι το φερόμενο Ισλαμικό κράτος έχει χρήματα για να χρηματοδοτεί τους οπαδούς του και διερωτώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέπτεται να κάνει κάτι για να κόψει την πρόσβαση του Ισλαμικού κράτους προς κονδύλια. Κύριος Μπρόχ, και εγώ έχω μια ερώτηση για τη Συρία. Ε, αναφέρθηκε σωστά ότι ε, η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, η πολιτική διαδικασία, πολύ σωστά όλα αυτά, Υπάρχει όμως αυτό το περίφημο θέμα των πληρεξουσίων, το proxy voice και κατά πόσον όλοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση. Σημείο 5 των συμπερασμάτων για τη Συρία, αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Εκεί αναφέρεται ότι η Ρωσία θα συνεργαστεί με Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία και τον Αραβικό Σύνδυσμο έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ειρηνική μετάβαση. Και έτσι λοιπόν το Συμβούλιο αποφασίζει να αναθέσει στην είπατε εκπρόσωπο να αναζητήσει ε, τρόπους για να υπάρχει πιο ε, επικοδομητική περιφερειακή συνεργασία. Κατ' εμέ αυτή είναι η πρόταση κλειδί των συμπερασμάτων και ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτής. Πολύ σωστά, πράγματι και καταλαβαίνω και την έννοια της ε, στασιμότητας και αυτής της σχετικής απογοήτευσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση στη Συρία. Δεν είναι προφανές, δεν προβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε τη Ρωσία, βλέπουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν ξέρω αν θα σας απογοητεύσω, αλλά εμείς δεν θα βομβαρδίσουμε. Εάν ε, το να προβληθούμε σημαίνει ότι θα πρέπει να βομβαρδίσουμε, θα σας απογοητεύσω. Εμεί δεν θα βομβαρδίσουμε. Η θέση μας είναι αυτή ε, η οποία μόλις ε, μας πέδειξε και ο Πρόεδρος. το έργο σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να μην προσελκύει τους πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες, αλλά περιμένω ε, τουλάχιστον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι περισσότερο. Ε, ε, εγώ και τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι προς αυτή την άγουσα θα πρέπει να επενδύσουμε. Τώρα αν θα προβληθεί αυτό δεν ξέρω. Σίγουρα ήταν αρκετά προβεβλημένο στο Ιράν και η συνάντηση που είχαμε σήμερα με την αντιπροσωπεία του Ιράν για το πώς μπορεί να ξεκινήσει η μετάβαση ε, στη Συρία ήταν πολύ σημαντική. Διότι εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε τους κατάλληλους ε, παίκτες ε, στη Συρία και πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία, κάποιος πρέπει να συζητήσει μαζί τους και κάποιος ο οποίος θα μπορεί να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνης τους ε, ή τουλάχιστον κάποιο βαθμό εμπιστοσύνης ε, και αυτός είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να συνομιλήσει μαζί τους και αυτό ακριβώς κάνουμε. Έγιναν τρει ή τέσσερι συναντήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Σαουδική Αραβία ε, τον περασμένο μήνα και με το Ιράν σήμερα το πρωί. Νομίζω εγώ και ανώτατοι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες ε, έχουμε ε, συζητήσει 6-7 ώρες με τους Ιρανούς ε, εταίρους μας και αυτούς που ήθελαν να μας επισκεφθούν. Το αν θα είναι στο πρωτοσέλιδο το New York Times αύριο δεν φαντάζομαι, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς και αυτό πρέπει να γίνει και ταυτόχρονα και εκ παραλίλου με αυτά που κάνετε μιστούρα στη Μόσχα και ε, μεθαύριο στην Ουάσιγκτον. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο διπλωματικού έργου το οποίο θα επιτρέψει να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Εμείς είμαστε δύναμη, αλλά πρέπει να διαδερματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι είμαστε ήπια δύναμη, αλλά πρέπει να είμαστε και μια ισχυρή δύναμη όταν υπάρχει ανάγκη να είμαστε ισχυροί και να επιδείξουμε την ισχύ μας δεν θεωρώ ότι το, Υπουργό, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θεωρεί ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε παράγον ασφαλείας και άμυνας στο θέατρο επιχειρήσεων της Συρίας. Ε, μπορεί να γίνει και σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων, να μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τους στρατιωτικούς μας ε, ε, μοχλούς ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κυρίως στο ανθρωπιστικό ζήτημα, ε, αυτό είναι άλλωστε κάτι που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό, και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να διοργανώσουμε διάσκεψη απαραίτητο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διοργανωθεί διάσκεψη ούτε ω Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ω Ηνωμένα Έθνη. Σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε το διπλωματικό και πολιτικό δίκτυο που θα μας επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας. Η διοργάνωση διάσκεψης είναι χρήσιμη όταν διαπιστώνουμε σαφώς τι συμπέρασμα μπορεί να προκύψει από μια διάσκεψη. Αλλιώς θα σπαταλήσουμε πολύ ενέργεια να διοργανώσουμε την ίδια τη διάσκεψη παρά να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Ιδίω δε σε αυτή την περίπτωση, όπου σαφέστατα θα πρέπει να συμμετέχουν οι διάφοροι παίκτε, οι διάφοροι παράγοντε ε, υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Εθνών και εντό του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, γιατί είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα για όλου όσοι συμμετέχουν, ώστε εγώ θεωρώ ότι το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είναι το μόνο υπό τη σκέπη του οποίου μπορούν όλοι να νιώσουν αρκετά άνετα και η ίδια η Συρία ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, Σαουδική Αραβία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι άλλοι ουσιαστικοί περιφερειακοί παράγοντες σίγουρα και οι Σύριοι που είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις περισσότερες επιφυλάξεις για τη συμμετοχή τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Επομένως η εντολή μας είναι αυτή ακριβώς, να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί διμερός ή πολυμερός σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη να ενθαρρύνει να ενεργοποιήσει, να διαμορφώσει, να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής προσέγγισης από τους βασικούς παράγοντες που συμμετέχουν και είμαι αισιόδοξη μετά από τη συνάντηση με τους Ιρανούς μας εταίρους σήμερα το πρωί ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Πολλοί από τους περιφερειακούς ε, παράγοντες διαπιστώνουν ή μπορεί να καταλήξουν να διαπιστώσουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη σύγκρουση και ε, σε αυτό εδράζεται και το διπλωματικό μας έργο. Όσον αφορά το ρόλο της Ρωσίας, ε, λυπάμαι που εξαρτώμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και νομίζω ότι το γεγονός ότι είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση σε καλύτερες πηγές από αυτές που έχουν οι δημοσιογράφοι. Σας ενθαρρυνώ λοιπόν να διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν εχθέ για το ρόλο της Ρωσίας. Μπορώ να σας τα διαβάσω κι εγώ αν θέλετε. Στην παράγραφο 10 λέει ότι οι πρόσφατες ε, στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας που πηγαίνουν πέραν ε, των επιθώσεων προς το Ισλαμικό κράτο και άλλων αποσχιστικών ομάδων είναι παραβίαση και πρέπει να σταματήσουν πάρα αυτά και όπως επίσης και η κλιμάκωση σε γειτονικές χώρες. Αυτή η κλιμάκωση σε στρατιωτικό επίπεδο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση και να αυξήσει τη ριζοσπαστικοποίηση. Στόχος μας είναι να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση και καλούμε τη Ρωσία να εντείνει την προσπάθειά τη ώστε να έχουμε μια ειρηνική επίλυση του ζητήματος και ζητούμε από τη Ρωσία να πιέσει για τη μείωση της βίας και την εφαρμογή μέτρων που θα δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στο Συριακό καθεστώς και όπως προβλέπει και το σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών 2131. Ζητώ λοιπόν, όπως θα έλεγαν και οι διπλωμάτες, να ε, εξετάσετε τα επίσημα έγγραφα και τις επίσημες δηλώσεις μας και όχι κάποια άρθρα που θα μπορούσε να γράψει ένας δημοσιογράφος στον τύπο, ορισμένες φορές με αυτά στοιχεία, ορισμένες φορές όμως με όχι τόσο ε, καλή πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν εμπορικέ ε, συναλλαγέ μεταξύ του Συριακού και του Λιβικού ζητήματος. Σε καμία περίπτωση ο πλήρης σεβασμός ε, και ε, και του Ικρανικού ζητήματος, συγγνώμη, ο πλήρης σεβασμός των συμφωνιών του Μίνσκ όσον αφορά την Ουκρανία είναι εκ των όνου κάνευ όρος. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη προσοχή στο θέμα αυτό, διότι η Ουκρανία, όπως και οι υπόλοιπε εταιρικέ σχέσεις ε, της Ανατολική Συνεργασίας, ήταν στην ημερήσια διάταξη και ο Ελμαρ Μπρόκ συμμετούχε και στην ε, ε, συζήτηση εκεί και νομίζω ότι το θεματολόγιο που έχουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων είναι αρκετά ισορροπημένο. Σίγουρα θα ξαναέρθει στο τραπέζι των συζητήσεων ε, τον ε, Νοέμβριο ε, ή τον Δεκέμβριο, γιατί πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει το θέμα των συμφωνιών του Μίνσκ μέχρι το τέλος του έτους. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Γκόμες ε, στην ανάγκη συντονισμού των κρατών μελών. Όταν είπα ότι είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην παρέμβει στρατιωτικά ούτε στη Συρία ούτε στην περίπτωση του Ιράκ, αυτό σημαίνει επιμένω ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε στρατιωτικές μας δυνατότητες σε άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε στον Διεθνή Συμμαχία κατά του φερόμενου Ισλαμικού κράτους. Το κάνουμε αυτό στο Ιράκ και στη Συρία. Το κάνουμε όμως με άλλα μέσα και όχι στρατιωτικά. Με πάση περιπτώσει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλα τα κράτη-μέλη μας συμμετέχουν με τον α ή με τον β τρόπο στη συμμαχία. Ορισμένα εξ αυτών δραστηριοποιούνται περισσότερο ε, σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στρατιωτικής φύσεως θέματα, άλλα σε άλλους τομείς. Στην προηγούμενη σταδιοδρομία μου πίεζα να υπάρχει ένα πλαίσιο, κοινό πλαίσιο για αυτές τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό εξακολουθεί να είναι η βάση. Ε, στις 15 Αυγούστου περασμένου έτους είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και αυτά έδωσαν σε όλα τα κρατημέλη ένα κοινό πλαίσιο γιατί χαιρέτησαν και στήριξαν τη συμβολή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στι στρατιωτικέ προσπάθειε προσπάθειες κατά του Ισλαμικού κράτους. Ως προς τον στρατιωτικό συντονισμό δραστηριοτήτων κάποιων κρατών μελών, ο συντονισμός αυτός ε, δεν πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας που δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πολλοί άλλοι παράγονες, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, όλοι συμμετέχουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήταν λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβαίνει σε στρατιωτικές ενέργειες χωρίς ε, να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν συμμετέχουν στη συμμαχία και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε πολύ καλά, εγώ ε, πάντα θέλω να υπάρχει συντονισμό των κρατομελών, έστω και στα στρατιωτικά. Αυτό θα επιθυμούσα και σε αυτή την περίπτωση. Αν δεν θεωρούσα ότι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή και σε αυτό το πλαίσιο δεν ενδείκνυται, δεν είναι αυτός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα στη Συρία, μισό λεπτό, έχω ακόμα να πω πολλά για την Τουρκία. Αυτά που σας είπα αφορούσαν στη συνεργασία, νομίζω εσείς κάνατε την ερώτηση, εσείς μάλιστα, η συνεργασία με αρχές και λαούς, οι πολίτες. Δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή όσο είναι τώρα. Βλέπω τα ερωτηματικά που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την όλη δυναμική που είχαν οι επιθέσεις και οι αντιδράσεις επ' αυτών. Θέλω να πω το εξή. Ανησυχώ ιδιαίτερα και πιστεύω ότι ο ρόλος μας πρέπει να είναι του να ενθαρρύνουμε πρώτα απ' όλα τη δημοκρατική εκλογική διαδικασία. Να συνεχιστεί αυτή, να λάβουν χώρα οι εκλογές στην 1η Νοεμβρίου ως προγραμματίζεται και αυτό σε ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει να ε, λάβει χώρα μια σωστή προεκλογική εκστρατεία, διαφανής, δίκαιη και όσο πιο ειρηνική γίνεται. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, εμείς δεν θα σταματήσουμε να ενταρρύνουμε τις τουρκικές αρχές, τα κόμματα και τους Τούρκους, τους πολίτες να επανέλθουν στην εσωτερική ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό είναι κλειδί για την Τουρκία, τους πολίτες της και την περιοχή. Ο ρόλος της Τουρκίας ε, στη μεταναστευτική κρίση και την κρίση των προσφύγων συζητήθηκε όχι μόνο χθες στους Υπουργούς Εξωτερικών, αλλά και στην ε, συνδιάσκεψη ψηλού επίπεδου των Βαλκανίων την περασμένη εβδομάδα παρούσης βεβαίως της Τουρκίας και προφανώς αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Να σας πω λοιπόν, κατανοώ πολύ καλά την πίεση που αισθανόμαστε όλοι στο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προσφύγων. Αυτό σε συνεργασία με την Τουρκία πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινή πρόκληση. Περίπλοκα όλα αυτά. Αλλά να πω επίσης ότι μόλις τελειώσαμε και να συζητάμε για τη Συρία και εφόσον το κλείσαμε αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικότερος διάλογος, ε, κοινή συνεργασία με την Τουρκία όχι μόνο για να διαχειριζόμαστε τις μεταναστευτικές ροές αλλά πρώτα απ' όλα συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο γιατί η Τουρκία αναμφισβήτητα είναι καθοριστικός παίκτη στην περιοχή και για τη Συριακή κρίση και για τις περιφερειακές ισορροπίες και εκτός αυτού είναι και μια χώρα με την οποία έτσι κι αλλιώς πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου για την περιφερειακή πολιτική. Ε, από την αρχή της θητείας μου είπα ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα για την Τουρκία που μπορούν να συζητηθούν. Νομίζω αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το πιο σημαντικό για την Τουρκία για να το συζητήσει μαζί μας είναι η εσωτερική ασφάλεια σε περιοχές ε, που έχουν άμεση σχέση με τις ε, αντιτρομοκρατικές επιθέσεις και όλα αυτά πάλι και σε σχέση ε, με την Συρία. Βεβαίως ε, και επαγγελματικές, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Πρέπει όμως ε, την Τουρκία να την αντιμετωπίζουμε όχι μόνο με κάποια ανανεωμένη ενέργεια όσον αφορά την ε, επανάληψη των συζητήσεων ε, για το θέμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην ξεχνάμε το περιφερειακό στοιχείο. Πολύ σημαντικό αυτό για μας. Τώρα, όσον αφορά, μάλλον να πω και κάτι άλλο, για τις ανατολικές ανατολικούς διαδρόμους των μεταναστευτικών ροών. Δεν σκεπτόμεθα οι αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τους διακινητές. Εμείς δίδουμε σημασία στην ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχει, υπάρχουν χώρες που ακολουθούν ε, την ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση και έτσι λοιπόν ε, μας δίνουν και διαφορετικά εργαλεία. Προφανώς τα χερσαία σύνορα είναι διαφορετικά από τα θαλάσσια. Έτσι λοιπόν οι δικές μας οι αποστολές έχουν στόχο να ενισχύσουν τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και αφορούν την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία. Και νομίζω ότι αν όλα αυτά τα αντιμετωπίσουμε με δυναμισμό θα αποδώσουν. Όσον αφορά τη Λιβύη και την επιχείρηση Σοφία. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Όταν πρότεινα το όνομα Σοφία, κάποιος είπε «Α, μα αυτό είναι όνομα γυναικείο» και εγώ έλεγα «Εντάξει, μια στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να έχει ένα γυναικείο όνομα, γιατί όχι». Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μικρό ανέκδοτο. Αυτή είναι, είναι το πρώτο ψήφισμα του ΟΗΕ, δεν ξέρω ποιος το ρώτησε αυτό. Ναι, αυτό ήταν ε, το πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ε, οπότε δεν ξέρω ακριβώς ε, σε ποια σύγχυση αναφερθήκατε όταν αναφερθήκατε στην, στο πρώτο ψήφισμα και το δεύτερο ψήφισμα. Για το πρώτο ψήφισμα μιλάω. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, για την εξαιρετική συνεργασία, όπως και την εξαιρετική συνεργασία των υπολείπων ε, κρατών μελών που είναι μέλη του Συμβουλίου, της, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καταφέραμε να έχουμε ε, μια πολύ, ένα πολύ καλό συντονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του ΟΗΕ, που είχε, αποτέλεσμα πολύ καλό, είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχουμε στο μυαλό μας να υπάρξει μια χερσαία επιχείρηση Όπω Όπως ξέρετε οι επιχειρήσεις έχουν διάφορες φάσεις. Ε, ακόμη είμαστε στο πρώτο τμήμα της δεύτερης φάσης. Έχουμε ακόμη το δεύτερο βήμα της δεύτερης φάσης, μετά μπορεί να περάσουμε σε τρίτο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα χερσαίων επιχειρήσεων στη Λιβύη για την ώρα ως τμήμα των επιχειρήσεών μας εκεί. Τρίτον, ε, το ότι διασώζονται λιγότεροι άνθρωποι. Εμείς με αυτήν την επιχείρηση που δεν έχει σκοπό όντως τη διάσωση αλλά το κάνει καταπολεμώντας ε, τους ε, λαθρέμπορους μεταναστών έχουμε διασώσει χιλιάδες ανθρώπους εκτός από αυτούς που έχει διασώσει Frontex με τις επιχειρήσεις τις αντίστοιχες που τις επιτρέπουν να κάνουν τη διάσωση. Δεν είμαι πάρα πολύ σε απόλυτους αριθμούς σίγουρη ότι όντως διασώθηκαν λιγότεροι. Εγώ νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν διασωθεί περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν. Ε, ε, ε όμως, ε, ήδη υπάρχει αποτέλεσμα. Ειδικότερα βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα στη διαδρομή αυτή ε, ίσως είναι το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησής μας. Αν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, ε, τι να σας πω. Ε, νομίζω ότι όχι. Το καλύτερο θα ήταν η Λιβύη να διαχειρίζεται τα σύνορα και να μπορεί να συνεργάζεται μαζί μας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κλπ. Αυτή τη στιγμή ε, αυτό είναι το αποτελεσματικό μέσο ε, που έχουμε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε οι εγκληματικές οργανώσεις να βγάζουν χρήματα από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή ε, δεν θέλουμε να βρουν εναλλακτικέ οδούς, ε, όχι, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ο αριθμός των συλλήψεων που έχουν γίνει και οι πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε κατά τις πρώτες φάσεις της επιχειρήσης είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές. Όσον αφορά τώρα το σύστημα αποτροπής το οποίο προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε για να μπορέσουμε να δυσκολέψουμε τους ε, εγκληματίες επειδή μιλάμε για επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό είναι το πρόβλημα ε, αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Επιμένω, συνεχίζω στη Λιβύη είναι πράγματι γεγονός ότι όλοι συμφωνούν με τη συμφωνία και μετά υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος αλλά το αναφέρατε αυτό, πράγματι ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι είναι είναι η τελευταία στιγμή κατά την οποία όλοι ε-, οι εταίροι μπορούν να καταλάβουν ότι το αλλά στο οποίο ε, αναφέρουν ε, εξουδεδιερώνει το αλλά κάποιων άλλον και το κοινό έδαφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη δυνατή εναλλακτική επιλογή που μπορούμε να έχουμε ως σημείο αφετηρίας. Αν καταφέρουμε να έχουμε ε, μία ε, κυβέρνηση. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ε, καταπληκτικό το αποτέλεσμα και παράδεισος από τη μια μέρα στην άλλη. Θα εξακολουθεί να είναι δύσκολη κατάσταση από απόψεως ασφαλείας, ειδικότερα κυρίως στην Τρίπολη. Αλλά, και αυτό είναι το δικό μου το αλλά, αν δεν καταλάβει ο κόσμος τη Λιβύη μάλλον να διορθώσω οι άνθρωποι που έχουν την πολιτική ευθύνη αρχίσουν να καταλάβουν, αν δεν αρχίσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να αφήσουν κατά μέρο τα αλά του και να μπορέσουν να βρουν κοινό έδαφο, θα συνεχίσει να ε, εκφυλίζεται η κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, ο λαό τη Λιβύη έχει κουραστεί με αυτόν τον πόλεμο και θέλει να βρει μία διέξοδο από την κατάσταση αυτή. Και ένα τμήμα τη δουλειά μόνο μπορεί να κάνει η διεθνή κοινότητα. Η βασική ευθύνη πρέπει να παραμείνει ε, στα χέρια των ε, ηθινών ε, ε, των υπευθύνων λήψη αποφάσεων ε, στη Λιβύη. Εμείς μπορούμε να είμαστε ένα εταίρο, αλλά η απόφαση πρέπει να είναι δική τους και αυτό είναι το σημείο της αφετηρίας μας. Δεν είναι δυνατόν εμείς να τους υποκαταστήσουμε. Ο ρόλος των περιφερειακών παικτών. Ναι, ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Όλοι, είτε η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλοι οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία του ελπίζω να συνεχίσει αυτό. Το SSRDDR, ναι, πράγματι κάνουμε μία προσπάθεια και ως προς αυτό, αλλά ε, είναι και πολλά ακόμη πράγματα τα οποία εξακολουθούμε να κάνουμε στη Λιβύη. Ίσως τα λέμε λιγότερα, ίσως για λόγους ασφαλείας, ε, όμως ε, έχουν να κάνουν με την υποστήριξη στην υπατερμοστία του ΟΗΕ εντό τη Λιβύη, ότι συνεχίζουμε να τους βοηθάμε και επίσης να υποστηρίζουμε και του Δήμου και τι κοινότητε. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα για τα οποία η Ένωση συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Λιβύη ακόμη και σε αυτέ τι δύσκολε ε, στιγμές. Όσον αφορά τώρα τη Λευκορωσία. Κοιτάξτε, αυτά δεν αποτέλεσαν τμήμα της χθεσινής μας ημερήσιας διάταξης. Ε, το συζητήσαμε κάπως. Ε, για τη Μέση Ανατολή μιλήσαμε για την εφαρμογή ε, κυρίως των αποφάσεων που έχουμε λάβει στο πλαίσιο του κουαρτέτου στη Νέα Υόρκη. Να προτείνουμε στα διάφορα μέρη συγκεκριμένα βήματα επιτόπου για να μπορέσουμε να να ανατρέψουμε τις πολύ αρνητικές εξελίξεις και να υπάρξουν κάποια θετικά, κάποιες θετικές εξελίξεις τουλάχιστον στην ε, Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό λόγω της κατάστασης ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Όμως το, προ... το δικό μου το μήνυμα προς ε, τον πρόεδρο Αμπάς και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου είναι ότι μην νομίζετε ότι το γεγονός ότι εκβιλίζεται η κατάσταση ασφαλείας είναι λόγος να μην ε, προσπαθήσουμε. Αντιθέτως είναι λόγος ε, να το κάνουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο επιγόντως. Όσον αφορά το θέμα της άρσης των κυρώσεων, ε, έφυγε ο συνάδελφός σας που έθεσε το θέμα, είναι ένα ε, ε, ερώτημα ε, πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τις εκλογές. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα, τα, τα πορίσματα των αποστολών παρατήρησης. Πρέπει να πω βέβαια ότι εμένα με ενθάρρυνε το να δω κατά τις τελευταίες εβδομάδες το γεγονός γεγονό ότι απελευθερώθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, όπω επίση και ότι οι εκλογέ έλαβαν ε, χώρα με ειρηνικό τρόπο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι μια χαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε την, ε, το τελικό πόρισμα. Οπότε από τη μία υπάρχει αναγνώριση των θετικών βημάτων και αυτό πιστεύω ότι συνιστά ένα θετικό μήνυμα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τη διενέργεια δημοκρατικών ε, διαδικασιών στη Λευκορωσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάτι ακόμη να πω ε, πριν από ένα χρόνο σας γνώρισα όλους, πρέπει να πω ότι έχω απολαύσει και έχω εκτιμήσει όλος ιδιαίτερος αυτή την πρώτη χρονιά συνεργασίας μαζί σας. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά Πολλά έχουμε ακόμη να κάνουμε, αλλά έχουμε ακόμη τέσσερα χρόνια κοινή εργασία. Έλμαρ, πραγματικά εκτιμώ όλο ιδιαίτερο τη συνεργασία και το συντονισμό μα. Ε, ε, ε, ίσως να το κάνουμε και καλύτερα από τι στρατιωτικέ δράσει των, των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ώρα. Πάντω ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία μα ω τώρα και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερω γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω αλλά ξέρεις Φεντερίκα, πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πάντοτε μπορούμε να γίνουμε καλύτερα. Ακόμη ελπίζω κατά τους επόμενους μήνες να μπορέσουμε να δούμε πώς θα βελτιωθούμε. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Και τώρα περνάμε στο διευρυμένο Προεδρείο.